για να αντιμετωπιστούν τα αποτελέσματα τα, όταν καταλάβουν τα αποτελέσματα αυτής της και τα κίνητα αυτής της επαναστάσεως που θα ολοκληρωθεί καλύτερα η κοινωνία της Ουκρανίας. Ευχαριστώ. Ακολουθεί η κυρία Κολάρσκα Μπομπίνσκα για δύο λεπτά. Dziękuję panie przewodniczący.